Χείρεψε η θέση του και τώρα λοιπόν να περάσουμε στο πρόγραμμα εργασίας. Η διάσκεψη του Προέδρου βάσει του άρθρου 169 του κανονισμού ενέκρινε την ημερήσια διάταξη. Mm. Και γι' αυτό λοιπόν προτείνω τις ε, εξής ε, αλλαγές στην ημερήσια διάταξη σύμφωνα με μετά από ε, συμφωνία με τις ε, ομάδες. Σε ό,τι αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, μετά από απόφαση του δικαστηρίου στις 16 ε, Δεκεμβρίου 2015, να μπει αυτό ως τέταρτο θέμα μετά τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για την διατραντική για τις διαπραγματεύσεις. Και έτσι λοιπόν η Ολομέλεια θα επεκταθεί μέχρι τις 12 το βράδυ. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά τις αλλαγές αυτές που προτείνονται. Ούτως λοιπόν θα τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη. Η ομάδα των Πρασίνων τώρα και οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζητούν η συζήτηση για το θέμα αυτό το οποίο σας ανέφερα να συνοδευτεί από ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί στην πρώτη ολομέλεια του Ιουνίου. Και για να ετυλογήσει το έτοιμο αυτό το λόγο έχει ο κύριος Λάμπερτς. Άση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποτίθεται ότι είναι ο θεματοφύλακος των συνθήκων ε, παραβιάζει αυτές τις συνταγές τουλάχιστον βάσει της γνωμοδότησης της νομικής μας υπηρεσίας η οποία λέει ότι δίχως αμφιβολία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει βάσει του άρθρου 266 ε, της συνθήκης της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σχετικό ψήφισμα διότι πιστεύω ότι είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να επανακαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τάξη, στην αποστολή της. Επομένως, ε, ε, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι το μέτρο δυσανάλογο, ε, εγώ θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, να έχουμε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην γίνει απλή συζήτηση μεταξύ μας, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει τα μέτρα που πρέπει. Ευχαριστώ. Υπέρ του αιτήματο το λόγο θα πάρει η κυρία Φαν Μπρέμπτ. Yes, thank um, Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζουμε το αίτημα των Πρασίνων. Όπως αναφέρατε, ήδη έκρινε το δικαστήριο σε σχέση με την αμφή Το των διατάξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο το ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει τελικά να υπάρχουν του ενδοκρινικού διαταράκτε αυστηροί στεγανοί κανόνε και να μην βασιζόμαστε κάποιο είδου ε, παράτυπη ε, αξιολόγηση επιπτώσεων αλλά σε επιστημονικά κριτήρια. Σα ευχαριστώ κύριε Φαμπρέν. Θέλει να πάρει κάποιο το λόγο κατά του αιτήματο αυτού. Δεν βλέπω να ζητά κανεί τον λόγο και γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε το αίτημα. Όποιο είναι υπέρ, παρακαλώ, τη ε, αίτηση αυτή. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνοδευτεί από ψήφισμα το οποίο και θα ψηφιστεί στην πρώτη ολομέλεια του Ιουνίου. Δεν ε, μεταβάλλεται η σημερινή ημερήσια διάταξη. Το ιωμά του ΕΝΕΦ ζήτησε μια δήλωση του Αντιπροέδρου είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτικής ασφαλείας για την μεταεκλογική κατάσταση στο Κονγκό να μπει σήμερα το απόγευμα στην ημερήξια διάταξη. Το λόγο έχει ο κύριος Αλιού. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση στην Μπραζαβίλ έχει καταστεί πάρα πολύ δύσκολη μετά από αυτό το παράνομο δημοψήφισμα, τόσο ώστε να παραταθεί η προεδρική θητεία που είναι πάνω από 3.000 και κατόπιν στις 20 Μαρτίου που είχαμε χαοτή κατάσταση. Είχαμε επίσης ε, σε όλη την περιοχή όπου κυριαρχεί η αντιπολίτευση έναν εντατικό ε, βομβαρδισμό και ε, έχουμε επίσης παρακολούθηση των ηγετών τη αντιπολίτευση και του στρατηγού Λοκό, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι πρόκειται για καταφανή καταπάτηση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ αμφιβολή εκεί πέρα η κατάσταση αφορά το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία. Θα πρέπει επομένω να δούμε την πραγματικότητα κατάματα και να κάνουμε για την Πρεζαβίλ μία συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ακόμα και το πιο ε, ανησυχητικό θέμα αυτής της χαόδους ε, ε, κατάστασης και το αίτημα της απόσυρσης του πρέσβη και της ανάκλησής του δημιουργία βεβαιότητα σε ένα πλαίσιο το οποίο περιγράφηκε πάρα πολύ καλά στην προηγούμενη παρέμβαση. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πάρα πολύ σοβαρής κατάστασης και γι' αυτό ακριβώς ε, πρέπει κατεπηγόντως να γίνει συζήτηση σε αυτό το κοινοβούλιο. Κύριος Μποργέτσι. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο κατά του αιτήματο. Όχι. Να ψηφίσουμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το αίτημα του κυρίου Άλιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το αίτημα. Και παραμένει λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, 40 μέλη βάση του άρθρου 113 παράγραφος 4 του κανονισμού τάχθηκαν κατά τι ε, διαδικασίε που ακολουθήθηκε για την έκθεση Κόβατσεφ σε ό,τι αφορά τι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 71η ε, Σύνοδο των ε, Ηνωμένων Εθνών. Και προτείνω λοιπόν αυτό να το κοιτάξουμε σε μελλοντική ε, συνεδρίαση. Υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Και περνάμε λοιπόν στην αυριανή ημερομηνία βάση του άρθρου 91 σε ό,τι αφορά την ασυλία της κυρίας τίφεται το θέμα αυτό και έτσι λοιπόν να σας πω ότι δεν πρόκειται για την έκθεση, για την στήλη της κυρίας Ρέγνερ. Όχι, είναι η συγγήτρια η κυρία Ρέγνερ για την... Ε, Τη έκθεση αυτή είναι λίγο σαφέ αυτό τα γερμανικά, λέει ο πρόεδρο. Η Γκουε ζήτησε μία δήλωση του Συμβουλίου για την υποτιθέμενη και εικαζόμενη διαπλοκή του Επιτρόπου Καλνιέτα σε περιπτώσεις διαφθοράς. Αυτό να μπει ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το λόγο λοιπόν έχει ο κύριος Μπενίτο Ζιλουάγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εκμεταλλεύτηκε τις ε, επαφές του για να δώσει την έγκριση ενός ε, κοιτάσματος ουρανίου στη ε, Σαλαμάνκα. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία είναι πολύ γνωστή του και εμφανίστηκε και στα Panama Papers. Υπάρχουν δύο έρευνες για διαφθορά οι οποίες αναφέρουν ότι ο κύριος Καλνιέτε είναι ένας από τους υπευθύνους και επίσης υπερψήφισε μία φορολογική αμνηστία όταν υπήρχε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Ε, πρόκειται λοιπόν για γεγονότα τα οποία αφορούν τον Επίτροπο για την Κλιματική Δράση και την Ενέργεια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι υπεύθυνο αν δεν δράσει ενώπιον αυτή τη κατάσταση. Όπω επίση θα είναι υπεύθυνη και η μεγάλη συμμαχία των ε, ε, σοσιαλιστών και του ΕΛΚ που επέτρεψαν αυτό το διορισμό και τον έκαναν μάλιστα και με άλλου διορισμούς. Εάν δεν ληφθούν μέτρα θα είναι ιδιαίτερα λυπηρό σχόλια εκτός μικροφώνου. Δεν αποφασίσαμε εμείς ε, ότι είναι αυτές οι υποθέσεις ε, πιθανής διαφθορές. Ε, θα είναι λυπηρό λοιπόν το γεγονός ότι το ΕΛΚ εξάγει ένα μοντέλο διαφθοράς και στην Ευρώπη. Το μοντέλο ενός κόμματος το οποίο παρανόμως χρηματοδοτείται για πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία. Έτσι είναι κυρίες και κύριοι. Ο Επίτροπος θα πρέπει να υπερασπίζεται τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες και θα πρέπει να έρθει εδώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δώσει εξηγήσει. Γιατί αλλιώς θα ζημιώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο. Κατά του αιτήματο. Κυρία Φαμπρέντ. Yes, Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του αιτήματο της ΓΚΟΕ σήμερα. Και όχι γιατί θεωρούμε το θέμα δεν είναι σοβαρό ή θα μπορούσε να καταστεί σοβαρό. Ούτε επειδή δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται πλήρες διαφάνεια σε τέτοια ζητήματα αλλά επειδή νομίζουμε ότι χρειάζεται και επειδή νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και για αυτού ακριβώ του λόγου θέλουμε νομίζουμε ότι χρειάζεται χρόνο μέχρι να αποφανθούμε. Θα πρέπει να δούμε το ζήτημα σε βάθο και κατόπιν να επανέλθουμε στην Ολομέλεια και να δούμε ποια είναι η πιο σωστή στρατηγική να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Προτιμούμε να έχει γίνει προηγουμένω μια συζήτηση ει βάθο στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Διαδικαστικό ζήτησα, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Διος Κανιέτε είναι ένας πολύ πρικισμένος ε, επίτροπος ε, και είδαμε τι έγινε μεταξύ άλλων και πώς ενήργησε στο COP21. Οπότε αυτή η δήλωση οικονομικών συμφερόντων πέρασε από την Επιτροπή και συνάδει με τον κώδικα διοντολογίας για τους επιτρόπους και καλύπτει όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητε και όλα τα οικονομικά συμφέροντα της ε, συζύγου όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την σύγκριση συμφερόντων. Οπότε νομίζω ότι υπήρξε εδώ ε, διαφάνεια αλλά για λόγους μικροπολιτικής η άκρα αριστερά από ευθύς εξ αρχής επιτίθεται στον Επίτροπο τον κύριο Κανιέτε και προσπαθεί με κάθε δυνατόν ε, μέσο να τον αμαυρώσει, ε, να τον υποβαθμίσει. Οπότε είμαστε κατά του αιτήματος. Ετέθησε, λοιπόν, έγινε το αίτημα αυτό και θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση για το αίτημα αυτό, όπως και ζητήθηκε. Έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Απορρίπτεται το αίτημα. Και έτσι παραμένει απαραλλακτή η ημερήσια διάταξη. Και τώρα να περάσουμε στις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Και το λόγο λοιπόν έχει ο Επίτροπος Άνζεπ. Αλλά αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Επίτροπε, θα περιμένετε λίγο.